Ο Κυρίες και κύριοι, ε, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, άρχεται η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι η ψηφοφορία για την αίτηση κατεπήγοντος πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού 1234 2007 ενιαίος κανονισμός ο ΚΟΑ με ε, τη θέσπιση ε, ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Ξαναδιαβάζω. Ε, πρόκειται για την θέση κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Η κυρία έχει, ο κύριος ε, Ντεκάστρο έχει το λόγο. Έχουμε ε, έχουμε ε, την ε, Επιτροπή Γεωργίας και ε, μία τόπο θέτηση της Επιτροπής Αλίας. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί φίλοι, Ξεκινάμε και πάλι ε, με τη συζήτηση του γαλακτοκομικού τομέα, ένα τομέα ο οποίος μας ανησυχεί πολύ και όπου η ε, γεωργοί ε, και οι αγρότες ε, ανησυχούν και εκδηλώνουν την ανησυχία τους. Έχουμε λοιπόν την υιοθέτηση της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ε, το γάλα είτε υγρό είτε σε σκόνη και έχουμε διατάξεις και για τα τυριά αλλά θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν και πρέπει να εξετάσουμε εάν θα πρέπει το άρθρο 186 της, ε, του, ε, του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ πρέπει να επεκταθεί και στο γάλα, δηλαδή να υπάρξει μία ε, διάταξη και ρύθμιση κατεπήγοντος χωρίς να περάσει από την κοινοβουλευτική εξέταση. και μία πρόταση της Επιτρόπου Fisher Bowl και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο